Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σας λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ γεμάτη μερίσια διάταξη σήμερα το πρωί. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Ως πρώτο θέμα της μερίσιας διάταξης είναι καταρχήν να την εγκρίνουμε. Η κυρία Αντρεάσεν έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Αντρεάσεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Παρακαλώ, προσθέστε στην ημερήσια διάταξή μας για σήμερα την συζήτηση ως τη συζήτηση για μένα που αναλαμβάνω τα καθήκοντα πρώτη αντιπρόεδρου. Και επίση θέλω να καταγγείλω τον κύριο Τζέσκαρο, ο οποίο ε, αλλίωσε τα αποτελέσματα τη εκλογή μα, αντιπρόεδρο. Λοιπόν, έχει κατεθεί αυτή η πρόταση της κυρίας Αντράσεν να αλλάξει η μερίσια διάταξη ε, και παρακαλώ να τοποθετηθούν το πολιτικές, πολιτικές ομάδες από αυτού. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Αντράσεν, ε, δεν θέλω να μπλεχτώ μέσα στην ε, διαμάχη ανάμεσα σας και τον κύριο Γκάιο, τον συνάδελφο, αλλά θέλω να επισημάνω ότι όλο αυτό δεν φέρνει τίποτα, δεν βοηθάει σε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω ε, να μην μπλεκόμαστε σε τέτοιου είδους ε, καταστάσεις. Ε, εσείς τώρα θέλετε να παραταθεί αυτή η ιστορία, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι καλή η ιδέα σας. Ο κύριος Γκάια, παρακαλώ, επί του θέματος. Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα, τοποθετήθηκα επ' αυτού στις συνεδρίες των συντονιστών και θα το ξανακάνω. Εγώ πράγματι ε, ξεκίνησα το σκεπτικό μου από λανθασμένα στοιχεία και κάπως έχασα και την ψυχραιμία μου και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη. Το γεγονός όμως ε, ότι επηρέασα τους ε, συναντέλφους, αυτό εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω. Από ό,τι θυμάμαι, Διάφορες πολιτικές ομάδες ε, τοποθετήθηκαν επί του θέματος ε, και είπαν ότι ε, θα υποστήριζαν την υποψηφιότητά σας και κυρίως διότι η αρχή don't για τις πολιτικές αυτές ομάδες θεωρείται πρώτης προτεραιότητας. Τώρα, κατά πόσον επηρέασα τη στάρφο κυρία Γκρέσλε με αυτά που είπα, δεν ξέρω, η ίδια η κυρία Γκρέσλε, Ίγκε, να απαντήσει από αυτού. Άλλος παρακαλώ, ο κύριος Μούλντα. Πάντοτε πρότειθα να συζητήσω τα πάντα, αλλά δεν νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι αυτή η επιπλέον ε, συζήτηση. Διεξήθη μυστική ψηφοφορία και το αποτέλεσμα προέκυψε και δεν ξέρω, δεν βλέπω εγώ να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ε, κατανοώ αυτό που ελέγχθη ως παράπονο καταγγελία, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιστραφεί το ε, από την ψηφοφορία. Ο πρόεδρος θέλει κάποιος άλλος. Ε, Το λόγο κύριε Μπάτον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, εγώ εκπλήσωμαι. Διότι δεν, καταλαβαίνω. Μου δώσανε εδώ πέρα τα σχετικά και φαντάζομαι θα γίνει ψηφοφορία. Τι να σα πω. Ε, κοιτάξτε στην άλλη Μπάρτονγκ, εξ όσων γνωρίζω, εσείς δεν είχατε δικαίωμα ψήφου, διότι η πολιτική, η πολιτική ομάδα εκπροσωπεί το ίδιο από κάποιον άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ε, κάναμε έλεγχο του καταλόγου ε, ποιοι μπορούν να ψηφίσουν και δικαιούνται ψήφου, ψήφο μόνο τα πλήρη μέλη ο συνάδελφός σας ε, ήταν παρόν, άρα δηλαδή ε, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε τη διαδικασία. Δεν ζήτησε κανείς άλλο το λόγο από τις ε, πολιτικές ομάδες. παρακαλώ λοιπόν τώρα να ψηφίσουμε για αυτό που πρότεινε η κυρία Ανδράσεν, δηλαδή κατά πόσον το θέμα το οποίο επιθυμεί θα προσθεθεί στη ημερήσια διάταξη όχι. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ της πρώτης κυρίας Ανδράσεν να ψηφίσουμε ανοιχτά. Όχι, καλύτερα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, ηλεκτρονικά. So, vote is open. Okay. So. Äh, λοιπόν, από τους μη εγγεγραμμένους μπορεί να ψηφίσει μόνο ένας. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν τώρα. Ψηφίζουμε παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ψήφισατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. 17 ψήφισαν, 15 ε, κατά, ένας ε, υπέρ και μία αποχή. Δεν αλλάζει λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Πολύ ωραία. Ε, πάμε τότε στην ημερήσια διάταξη, την οποία εγκρίνουμε και ως έχει. Άλλες προτάσεις για την ημερήσια διάταξη, από ό,τι βλέπω όχι. Κατόπιν τούτου εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών και εδώ σας παραπέμπουμε στα σχετικά πρακτικά. Από ό,τι βλέπω ε, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, γκρίνεται και το θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, το σημείο υπαριθμών 4. Και συγκεκριμένα πρόκειται για τον ορισμό ενός μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας παραπέμψω στην ακρόαση που έλαβε χώρα στην Επιτροπή μας ε, και καλωσορίζω τον κύριο του Μουγκουρούζα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Στη διαδικασία που προβλέπετε, ο υποψήφιος, ο κύριος Μουγκουρούζα, ε, θα συστηθεί, θα παρουσιάσει τον εαυτό του. Ε, μετά η συγγήτρια θα κάνει κάποιες ερωτήσεις και κατόπιν, αφού ακούσουμε την απάντησή του, θα μπορούν και οι άλλοι συνάδελφοι να υποβάλουν ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω θερμά και να σας παρακαλέσω να λάβετε το λόγο. Παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη το μικρόφωνο που είναι αριστερά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτέ. Μεγάλη μου χαρά, εμφανίζομαι εδώ ε, στην ε, Επιτροπή του ε, Ελέγχου Προπολογισμού εκπροσωπώντας ε, την, την Ισπανία για την υποψηφιότητα αυτή όσον αφορά δηλαδή το ελληνικό συνέδριο. Όλοι έχετε το βιογραφικό μου και επίση τι απαντήσει μου. Οπότε θα πρέπει για λίγα λεπτά να σα πω κάποια σημεία από την σταδιοδρομία μου και από την παιδεία μου που θεωρώ ότι σχετίζονται άμεσα με τα ενδεχόμενα καθηκοντά μου στο ελεγκτικό συνέδριο. Όταν ολοκληρώσα τις σπουδές μου, σπούδασα νομική, ε, έγινα, αφού πέρασα έναν διαγωνισμό, επιθεωρητής οικονομικών για το Ισπανικό κράτος. Από τότε ε, ακριβώς ε, ασχολούμαι το Υπουργείο Οικονομικών και ως επιθεωρητής εξειδικεύτηκα στα φορολογικά και όσον αφορά τους ε, οικονομικούς ελέγχους. Και έτσι επομένως απέκτησα μια σφαιρική άποψη από τα θέματα ε, τα δημοσιονομικά και τα νομικά. Ε, τα καθηγόντά μου στο Υπουργείο Οικονομικών αφορούσαν την εκτέλεση της φορολογικής νομοθεσίας, την εφαρμογή του φορολογικού δικαίου και κυρίως όσον αφορά τις εταιρείες, τα λογιστικά, Οτι οτιδήποτε έχει σχέση επομένως με αυτά, αυτές τις ε, υποθέσεις και ε, επομένως έτσι μπόρεσα να μάθω σε βάθος τι γίνεται όσον αφορά ε, το, το, το, τη φορολογική πολιτική. Οπότε και μπόρεσα να σπουδάσω και στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια υποτροφία του Υπουργείου σε, στο Εθνικό Ευθύνη της Αμερικής επίσης ε, είμαι και μέλος του οικονομικού διοικητικού δικαστηρίου της χώρας που επιλύει διαφορές φορολογουμένων κατά του κράτους. Το 1996 πήγα στο ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού της χώρας. Πρώτα-πρώτα διευθυντής για οικονομικά και κοινωνικά θέματα και κατόπιν διευθυντής της ε, υπηρεσίας επί του προπολογισμού. Οπότε μπόρεσα να ε, συμβάλλω κι εγώ όσον αφορά το τι αποφάσιζε ο Πρωθυπουργό για τη δημοσιονομική πολιτική και για την φορολογική. Ακριβώς τότε λίγο πριν ε, θεσπιστεί το ευρώ η Ισπανική κυβέρνηση, το Ισπανικό κράτο προσπαθούσε να ε, συμμορφωθεί με τα κριτήρια του Μάστριχτ και επίση να μπορέσει να φέρει μια εξυγίανση στη δημοσιογραφία τη χώρα. Κατά την ίδια περίοδο επίση συμμετέσχουν στην ε, προπαρασκευή και διαπραγμάτευση ε, που έκανε η Ισπανία για τι δημοσιονομικές προοπτικέ περίοδο 2000 και 2006. Και έτσι, έτσι απέκτησα μια καλύτερη οπτική των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών. Επίσης, 2000 και 2002 ε, ήμουν ε, υπουργό τηλεπικοινωνιών και της κοινωνίας της πληροφορίας. Από το 2004 είμαι βουλευτής. Και εκεί ασχολούμαι με τα δημοσιονομικά, τα οικονομικά του κράτους γενικότερα και συμμετέχω στην αντίστοιχη επιτροπή της Ισπανικής Βουλής 25 χρόνια. επομένω έχω υπηρετήσει τα δημόσια πράγματα σε, σε ψηλό επίπεδο και στη δημόσια αλλά και βουλευτής. Στο Υπουργείο Οικονομικών και επομένω διάφορου άλλου ρόλου ρόλους έχω αναλάβει όσον αφορά τα δημοσιονομικά ε, δαπάνες και έσοδα. Και πιστεύω ότι επί τη βάση της εκπαίδευσή μου αλλά και της επαγγελματική μου εμπειρία θα μπορέσω αποτελεσματικά να βοηθήσω όσον αφορά τα καθήκοντα αυτά, τα οποία πρέπει να ε, αναλάβει κανεί στα πλαίσια του ελεγκτικού συνεδρίου. Εν κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα πω μια σύντομη σκέψη μου όσον αφορά το πόσο σημαντικό είναι το ελεγκτικό συνέδριο ε, όσον αφορά την σημερινή συγκυρία της οικονομικής ε, και δημοσιονομικής ε, κρίσης. Υπάρχει σπάνιες όσον αφορά τους πόρους. Οι πολίτες ελπίζουν και απαιτούν όσον αφορά τη σχέση τους με το δημόσιο. Επομένως χρειάζεται πάρα πολύ σημαντική διαχείριση, χρειάζονται οικονομίες, αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει όμως όλα αυτά να γίνουν με διαφάνεια, υπευθυνότητα, απόδοση λογαριασμών και συνεχή αξιολόγηση της διαχείρισης αλλά και της ε, ασκουμένης το ελληνικό συνέδριο είναι ελεγκτής, εξωτερικός και ανεξάρτητος. Οπότε, νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει όσον αφορά την ανάκτηση της ε, εμπιστοσύνης των πολιτών και επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των ε, χρημάτων και πολιτικών της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να απαντήσω σε τυχόν ερώτηση. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Μουκούρθο για την εισήγησή σας και τώρα δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ που είναι η εισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε κύριε Μουγρούθα στην Επιτροπή μας. Είναι, είσαστε λίγο στριμωγμένος, οπότε δεν σας ζηλεύω για τη θέση σας, γιατί για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο έχουμε πρόταση κυβερνητική κάποιου που έχει την δική σας διαδρομή έγκριση από την Ολομέλεια. Ε, αυτό έχετε αυτό το αμερόληπτο προφίλ και επομένως όσον αφορά τα, την ουσία του πράγματος ε, νομίζω ότι μπορείτε εσείς να ενταχθείτε στον εξάρτητο αυτό όργανο το ελεγκτικό συνέδριο. Ακριβώ όπως ισχύει και στις χώρες μας. Ε, όμως, είχαμε την απόσταση της υποψηφιότητα από, το, ε, από την Ισπανία και μετά ξανακατεβήκατε υποψήφιο. Και συγκρίνουμε τα προσόντα σα την ηλικία σα με, σε σχέση με τον προκάτοχο. Δεν, δεν αφήσουμε τίποτα από όλα αυτά, όμως ε, μένει ένα ερωτηματικό. Το ερωτηματικό είναι η αμεροληψία, η ανεξαρτησία σας. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί έγινε αυτή η αλλαγή και σε σχέση με την ε, ενδυνάμει ανεξαρτησία σας. Είναι πάρα πολύ βασικό το να είστε ανεξάρτητος. Είπατε ότι είσαστε μέλος του Προεδρείου του Λαϊκού Κόμματος. Καλά, όλοι εδώ είμαστε βουλευτές, έχουμε σχέση με κάποιο κόμμα. Εσείς όμως είσαστε μέλος του Προεδρείου του Λαϊκού Κόμματος και υποθέτω ότι ο μισός μισθός σας από εκεί προέρχεται. Βέβαια, και ο προκάτοχος συμμετέσχε σε κομματικό think tank. Αλλά τον είχαμε ρωτήσει σχετικά και εκείνον. Εγώ τον είχα ρωτήσει. Για πέστε μας επομένω, δεν θέλουμε να είστε ανεξάρτητο. Τι λέτε. Επίσης, εσείς έχετε συμβάλει πάρα πολύ στα δύο τελευταία προεκλογικά προγράμματα του Λαϊκού κόμματο της Ισπανίας. Είσαστε επομένω. όχι απλώς μέλος του Προεδρείου, αλλά σα είχε αναθέσει το κόμμα σα να συντάξετε αυτά τα προεκλογικά προγράμματα. Επίσης, σε σχέση με αυτό που μας είπατε εσείς για τα δημοσιομικά με το οποία έχετε ασχοληθεί, έχουμε την αλλαγή μεταξύ του καθηγητή Βαρέα και ημών. Εκείνος ήταν ο εμπειρογνώμων που προετοίμασε την ε, είσοδο της Ισπανίας στο ευρώ. Είχε θεωρήσει επομένω η κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματο να κατεβάσει τον καθηγητή εκείνο. Όμω τώρα έγινε η αλλαγή και κατεβάζουν εσά ω υποψήφιο, που είσαστε λιγότερο ανεξάρτητο. Μα είπατε ότι έχετε κάνει στον φαντηγή των δημοσιονομικών, το, το, πρόγραμμα Redes δίκτυα στην Ισπανία, ασχοληθήκατε με όλα αυτά και όμως κάποια στιγμή η τράπεζα BBVA είχε πει ότι δεν είχε όλα τα στοιχεία σε σχέση με τη δική σας διαχείριση. Δεν δίνατε εσείς δηλαδή τα στοιχεία στην τράπεζα όσον αφορά επομένως τα τότε καθήκοντά σας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα διαφάνειας. Επίσης, κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Ε, στο τέλος του ερωτηματολογίου πάντοτε το Κοινοβούλιο ρωτά τι θα γίνει, τι θα κάνετε εάν απορριφθεί η υποψηφιότητά σας. Το Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο υποχρεούται να μια, μια που είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών, θέλουμε επομένως να γίνετε σεβαστή, να λαμβάνετε υπόψη η γνώμη μα. Εάν επομένως εμείς είμαι αρνητικοί θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σα. Όμω η απάντηση που δίνετε εδώ δεν μα ικανοποιεί. Ενώ τα είχε πει πιο ξεκάθαρα ο προηγούμενος υποψήφιος. Επίση ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε εκείνη να αναθεωρήσει την υποψηφιότητά σα σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης. Όμω πέστε μας, μπορείτε εσείς να μας διαβεβαιώσετε ότι θα αποδεχθείτε την αρνητική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Συγητρία, ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ για τις ερωτήσεις που θέσατε στον υποψήφιο και θα τον παρακαλέσω να απαντήσει ευθύ αμέσω στι ερωτήσει αυτέ. ερωτήσεις αυτές. Έχετε το λόγο κύριε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ένα σωρό ερωτήσει μου υποβλήθηκαν από την κυρία Γιάλα Σέντερ. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Όσο γίνεται. Εάν κάτι δεν καταστεί σαφές, ξαναρωτάτε. Από ό,τι κατάλαβα, στην αρχή αναφερθήκατε στο κατά πόσον είμαι ανεξάρτητος ως μέλος ή υποψήφιος για το ελληνικό συνέδριο. Η δέσμευσή μου είναι μόνο μία. δέσμευση προς το ελληνικό συνέδριο Γι' αυτό και αποκλειστικά θα ασχολούμαι μετά του ελεγκτικού συνεδρίου, όπως απαιτείται από το καταστατικό του και όπως λέει και η συνθήκη. Αυτό για μένα είναι σαφές. Δεσμεύομαι προ τούτο. Ανεξαρτησία. Στη δική μου περίπτωση μπορείτε να διαπιστώσετε την ανεξαρτησία μου μέσω της ε, εκπαίδευσης, παιδείας, σταδιοδρομίας μου είναι άκρος τεχνικά και τεχνοκρατικά τα καθήκοντα κάποιου στο ελεγκτικό συνέδριο. Κανείς έχει ως αρρωγούς τις ίδιες τις υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου μόνο. Οπότε, οι αρμοδιότητες ρυθμίζονται από το καταστατικό του ελληνικού συνεδρίου και παρέχονται όλες οι εγγύσεις της ανεξαρτησίας. Και εγώ επίσης έχω διατελέσει επιθεωρητής οικονομικών για το Ισπανικό κράτος. Εκτέλεση και εφαρμογή του προπολογισμού ήταν και αυτό ένα από τα καθήκοντά μου και νομίζω ότι βάσει αυτή τη διαδρομή μου όλα αυτά δείχνουν την ανεξαρτησία μου. Δεύτερον, ρωτήσατε τι θα γίνει αν τι, τι, τι, έγινε με, με αυτή την αλλαγή της υποψηφιότητας. Ξέρω το, το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο διχάζει αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτε γιατί τα έκανε αυτά η Ισπανική κυβέρνηση. Εδώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σας πω τη γνώμη μου και για κάποιον άλλο, όπως εσείς αναφερθήκατε προηγουμένως, στον καθηγητή, καθηγητή Κορώνα. Είναι αξιοσέβαστος και γνωριζόμαστε εδώ και μία εικοσαετία. Οπότε παρακαλώ να με κρίνετε επί τη βάση της ε, παιδείας μου και της σταδιοδρομίας μου. Αυτά είναι τα κριτήρια και όχι κάτι το οποίο εξαρτάται και σχετίζεται με κάποιο άλλο πρόσωπο. Τώρα όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή του Λαϊκού κόμματο στην Ισπανία. Η συμμετοχή μου εκεί δεν είναι μυστικό, το έχω πει και στο ερωτηματολόγιο και ξεκάθαρα νομίζω ότι απήντησα στο ερωτηματολόγιο. Υπήρχε απευθεία άμεσο ερώτημα το οποίο τίθετο και εγώ απήντησα και σα είπα ότι προβλέπονται όλα αυτά και από το καταστατικό και καλύπτουν το καταστατικό του Ελληνικού Συνεδρίου. Και εννοείται ότι όταν ε, αναλάβω τη θέση μου στο Ελληνικό Συνέδριο θα παραιτηθώ από κάθε θέση που έχω στο Λαϊκό Κόμμα και επίσης θα παραιτηθώ και από, την, το βουλευτικό μου αξίωμα. γνώσεις, ε, εμπειρία, όλα αυτά θα τεθούν στην υπηρεσία του Ελληνικού συνεδρίου ακριβώς όπως ε, προϋποθέτουν τα καθήκοντα για να της αποστολής μου εκεί. Τώρα, όσον αφορά την, ε, το, πολιτικό ίδρυμα στο, του οποίου ήμουν γενικός γραμματέας, αυτό το ΦΑΕΣ, μεταξύ το 2000 και το 2004, ε, είχα αυτή τη θέση. Οργάνωσε αυτό το νέο ίδρυμα και από το 2004 είμαι απλό μέλος. και υπάρχει άλλος γενικός γραμματέας και εκτελεστικός διευθυντής. Επίσης, έχω διατελέσει διευθυντής του, της υπηρεσίας για τα δημοσιονομικά από το 1998 μέχρι το 2000. Επρόκειτο για υπηρεσία που ε, βοηθούσε τον Πρωθυπουργό και επίσης ε, συνεργάστηκα με τον καθηγητή Μπαρέα. Καθηγητής, ε, σύμβουλος, υπουργός, ε, άνθρωπος υψής του κύρου στη χώρα μας και ε, τότε περάσαμε από μια αναδιοργάνωση των υπηρεσιών που είναι αρρωγή του Πρωθυπουργού στην ιδέα του καθηκόντων του. Εγώ ασχολήθηκα λοιπόν με τα οικονομικά και τα κοινωνικά και υπήρχε και πιο εξειδικευμένη υπηρεσία υπό τον ε, καθηγητή Μπαρέα. Όπως ξέρετε ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικά, σημαντική η συμβολή του τότε για την εξηγήση των οικονομικών από το 1996 και μετά και καταφέραμε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την είσοδο στο ευρώ. Μέχρι το 98 γίνανε αυτά. Επομένω πρόκειται επίσης για πάρα πολύ σημαντική σταδιοδρομία, η σταδιοδρομία του κυρίου Μπαρέα και ε, σημαντικός πανεπιστημιακός θεωρείται. Κάποια στιγμή επομένω είχαμε αναδιοργάνωση τη υπηρεσία και ανέλαβα εγώ τα καθηγητά του καθηγητού Μπαρέα. Παρακάτω. με ρωτήσατε τι γίνεται όσον αφορά τα καθηκοντά μου στο Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας. Από το έτος 2000 έγινε και εκεί αναδιοργάνωση στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κυβερνητικής και για πρώτη φορά συγκροτήθηκε ένα τέτοιο Υπουργείο το οποίο είχε ως χαρτοφυλάκιο όχι μόνο τα ρυθμιστικά για ίντερνετ και τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικά, αλλά είχαμε και την αποστολή να συντονίσουμε. τον τρόπο οριζόντιο τη δράση όλων των Υπουργείων σε σχέση με την κοινωνία της Οριζόντιο για όλους τους φορείς, όλα τα Υπουργεία όλη τη διοίκηση. Υγεία, παιδεία, ΜΜΕ. Ό,τι εσείς με γιονές πληροφορία σε όλους αυτούς τους τομείς. Οπότε, εγώ είχα λάβει τον συντονισμό. Χρησιμοποίησαμε τους πόρους που είχαν διατεθεί για τους σκόπους αυτούς. Βέβαια, δεν, μπορούσαμε κάθε φορά να κάνουμε όλη τη δουλειά εμείς γιατί για, για, το, για, για, το, πρόγραμμα, για το όραμα, η ηλεκτρονική η e-health, υπήρχε το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως, είναι αλήθεια ότι γινόταν η πολιτική ζήμωση και όντως, όπως λέγατε και εσείς, φτάσαμε σε εκτέλεση 182% του προπολογισμού. Και όντω και εγώ έχω θεωρήσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Όμως, αυτό το οποίο τότε καταφέραμε είναι να υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία και συνεχίστηκε, έστω και αν βαφτίστηκε αλλιώ. το για το οποίο είναι σύνηθε το κάνουν οι κυβερνήσει Νομίζω ότι στρατηγική εκείνη την οποία εγώ εσχεδίασα ήταν και παραμένει πάρα πολύ αποτελεσματική. Βέβαια όσο γίνεται πιο σημαντική η κοινωνία πληροφορία τόσο περισσότερο απαιτείται μια τέτοια συγκρότηση της υπηρεσίας σαν και εκείνη. Τώρα, το άλλο θέμα τη συμμετοχή μου στον ε, συντονισμό των ε, προεκλογικών προγραμμάτων του κόμματός μου. Από το 2004 έγινα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τότε εκτός από τα άλλα μου καθήκοντα στις κοινωνικές επιτροπές ή, ε, ήμουν επίσης και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανέλαβε επομένω ε, σε, σε, τρει περιπτώσει ανέλαβα τα προεκλογικά προγράμματα του κόμματο. Μου ανέθεσαν επομένω τον συντονισμό των προεκλογικών ε, προγραμμάτων. Πρώτα-πρώτα αυτό έγινε το 2004. Και το 2011 επίσης ε, είχα αναλάβει τέτοιο συντονισμό ένα πρόγραμμα πλαίσιο. Έτσι πλαισιώθηκαν στις ε, τοπικές και περιφερειακές εκλογές υποψηφοί του κόμματός μου, αλλά είχαν λάβει και το πρόγραμμα για τις βουλευτικές εκλογές. Τώρα να σας πω μια σκέψη μου γεννήθηκε ότι ένα προεκλογικό πρόγραμμα έχει πολλές πτυχές. Είναι όργανο, μέσο πολιτικής επικοινωνίας. Όμως προϋποθέτει σφαιρική γνώση των πολιτικών της κάθε κυβέρνησης. Νομίζω σας εκάλυψα στις ερωτήσεις σας. Ε, ευχαριστώ κύριε Τομιμού Κορόσα. Έχουμε άλλωστε ακόμη έναν αριθμό ερωτήσεων και επί της διαδικασίας θα προτείνω να βάλουμε όριο στο χρόνο αγορεύσεως. Αλλά υπάρχει μια σύντομη συμπληρωματική ερώτηση της κυρίας Αγιά Σέντερ. Ναι. Συγγνώμη Πρόεδρε, συμπληρωματική ερώτηση. Δεν είναι συμπληρωματική τόσο πολύ, αλλά δεν μου απήντησε ο κύριος Μουγκρούθα. Το τελευταίο που είπα, τι θα κάνει εάν το Κοινοβούλιο δεν τον περιβάλλει με την εμπιστοσύνη. Και άρα απορρίψει την υποψηφιότητά του. Μουγκρούθ. Σε σχέση με την τελευταία σα αυτή ερώτηση και του ερωτολογίου, είχα πει ακριβώ ότι ελπίζω να με περιβάλλετε με την εμπιστοσύνη μα σε επί τη βάση της αδειοδρομία μου και το ότι θα έχω την εξαρτησία που επιβάλλει η συνθήκη. Επίση, είμαι πεπισμένο ότι οι σχέσει μεταξύ ελεγκτικού Συνεδρίου και Κοινοβουλίου θα χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη και συνεχή διάλογο. Οπότε, ε, εάν έχετε εσεί αρνητική γνώμη όσον αφορά τι ικανότητέ μου, τι επαγγελματικέ, θα ζητούσα από την Ισπανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την ε, υποψηφιότητά μου. Νομίζω ότι είμαι σαφή. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να αναλάβω εγώ τα καθήκοντά μου στο Ελληνικό Συνέδριο να με υποστηρίξει το Κοινοβούλιο. Έχει νόημα η διαβούλευση που γίνεται τώρα. Άρα και εσείς θα πρέπει να κρίνετε εάν η εκάστοτε υποψήφοι είναι κατάλληλοι για τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται. Αυτό είναι και ο δικό σα ρόλο, οπότε γι' αυτό είπα και αυτό που είπα, ότι θα ζητήσω αναθεώρηση τη ψηφιότητό μου σε αρνητική περίπτωση, εάν ε, δηλαδή θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι δεν συγκεντρώνει σε πρώτες προϋποθέσεις. Θα ζητήσω η κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της, ξαναλέει ο κ. Μουγκουρούθ. Όμως, δεν είμαι εις θέση να σας πω άμεσα ότι θα παρετηθώ, γιατί δεν πρόκειται εδώ περί υποψηφιότητα σε κάποιο διαγωνισμό. Η υποψηφιότητά μου ολοκληρώθηκε κατόπιν κάποιε διαδικασίε και είναι η ψήσιμη υποψηφιότητα τη Ισπανική κυβέρνηση. Θεωρώ πάντως απαραίτητο το να με υποστηρίξει, το να έχω την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου για να λάβω τις αρμοδιότητες μου, διότι η χώρα από την οποία προέρχομαι υπάρχει μια παράδοση εξωτερικού ελέγχου όπου η, το κοινοβούλιο ορίζει τα μέλη του Ισπανικού Ελληνικού Συνεδρίου. Äh, Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ακολουθούν οι εξής συνάδελφοι. Ότις, Γκάιος, Κυλακάκης και Και θα προτείνω να κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων 1,5 λεπτό για τις ερωτήσεις, 3 λεπτά για τις απαντήσεις. Ελπίζω να μπορέσουμε όλοι να τηρήσουμε λίγο πολύ αυτό το χρονικό όριο. Ευχαριστώ. Κύριο Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν θέσω την ερώτησή μου, θα κάνω μια παρατήρηση σχετικά με την παρέμβαση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, η οποία στο 80% της παρεμβάσεώς της στην ουσία έκανε ε, δίκη προθέσεων ε, του υποψηφίου. Στην πραγματικότητα εσείς δεν είστε ανεξάρτητοι, διότι είστε μέλος ε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας, Είναι ασκείτε πολιτική. Θα μπορούσατε όμως για το ντοσχέ αυτό να υποβάλλετε την θέση σας στον εισηγητή, διότι βρίσκεται σε σύγκρουση Συμφέροντων. Κατάλαβαν οι Ισπανοί Σοσιαλιστές ότι χάσανε τις εκλογές. Ίσως και εμείς να τις χάσουμε. Ελπίζω όχι. Πιστεύω πως όχι. Γιατί θα ήταν, θα ήταν άσχημο νέο. Αλλά πρέπει να παίζει κανείς σωστά με τους κανόνες. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία άλλαξε. Λυπούμε πολύ που η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού πολιτικοποιεί εν πάση περιπτώσει μια υπόθεση που έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα. Εσείς κύριε Τομέ Μουγκουρούζα, έχω μια ερώτηση να σας κάνω. Έχετε προ προετοιμαστεί βέβαια για την ακροασή σας. Γνωρίζετε ότι εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού προωθούμε την ιδέα να υπογράφουν αρχή κατών και κυβερνήσεων δήλωση αξιοπιστίας. Εάν θα είστε μέλος, εάν θα γίνετε μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, πώς βλέπετε τις σχέσεις που μπορεί να διατηρείτε με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Έχω προτείνει μια ιδέα που ακόμα δεν υποστηρίζεται από μεγάλη πλειοψηφία, αλλά πάντως είναι μια ιδέα στον έλεγχο δηλαδή και ιδίω της επιμερισμένης περισμένου ελέγχου, δηλαδή των κονδυλίων που διαχειριζόμαστε μαζί με τις ε, χώρες μέλη, να γίνεται κοινή, ε, να γίνεται συνεργασία μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευρωπαϊκού με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Έχετε βέβαια στην εμπειρία σας και πολλά χρόνια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Ισπανικό και γνωρίζετε τον τρόπο που λειτουργεί ο υπεψήφιος Ο πρόεδρος μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Τι. Παρακαλώ, απαντήστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω και όταν το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο ασκεί έναν ε, έλεγχο επί του κοινωτικού προϋπολογισμού και επί της εκτέλεσης των κοινωνικών προϋπολογισμών, των κοινωνικών πολιτικών, ως επιτοπλίστων η διαχείριση και ο έλεγχος γίνεται επί κάποιων διαδικασιών και κάποιων δαπανών που πρακτικά ε, έχουν τελεστεί από κάποιες εθνικές αρχές και φορείς. Επίσης, πολλές φορές ε, καλούνται τα εθνικά λεκτικά συνέδρια να συνεπικουρήσουν. Πολλές φορές, επομένως, υπάρχουν εδώ πέρα συντρέφουσες ομοδιότητες και αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και ε, τη δράση μας με τα Εθνικά Ελληνικά Συνέδρια, ούτως ώστε να μην έχουμε επικαλύψεις. Και επίσης να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες ε, κοινέ κινήσεις, ούτως ώστε να είναι δυνατόν κάποιο θεσμικό όργανο να στηρίζεται ε, στο έργο κάποιου άλλου θεσμικού οργάνου και όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο ή και εξωτερικό, ως, ανάλογα με το θεσμικό όργανο, θεωρώ ότι ε, βεβαίω είναι μια δύσκολη δουλειά και δαπανηρή πολλές φορές επομένως ε, και επίπονη θα πρέπει βεβαίω όλη αυτή η διαδικασία να καταστεί αποτελεσματική Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει φυσικά αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινέ διαδικασίε, κοινοί κανόνε για να γίνουν κοινοί έλεγχοι. Μέχρι τώρα αυτή καταβάλει προσπάθεια προ τούτο από τα έλεγχτικα συνέδρια. Και αυτό ισχύει για, όλα, για όλους τους ελληνικούς οργανισμούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Ριβελίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα και εγώ να κάνω μία σκέψη. Την εξή, ότι <clears throat> το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάψει να είναι υποκριτικό. Να κοιτάει την ουσία και όχι τόσο τον τύπο. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε προκατηλημένοι. Εμείς καλούμεθα να αποφασίσουμε. Πρέπει λοιπόν να διερωτηθούμε κατά πόσον ο υποψήφιος τον οποίο αξιολογούμε σήμερα, κατά πόσον έχει τις τεχνικές γνώσεις, κατά πόσον ο υποψήφιος είναι τίμιος, ε, αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τη σκέψη ότι αν ανήκει σε ένα κόμμα ή σε άλλο γιατί για μένα είναι διάφορα αν κάποιο είναι οπαδό τη Ρεάλ Μαντρίτη ή τη Μπαρσελόνα. Εμένα με ενδιαφέρει κατά πόσον ο υποψήφιο έχει την τεχνογνωσία να κάνει τη δουλειά του. Μα κανεί δεν είναι απόλυτα ουδέτερο. Και αν καλούμε ε, να κρίνω έναν υποψήφιο με βάση το ποδόσφαιρο, ε, και εκεί εμένα με ενδιαφέρει αν τεχνικά είναι προετοιμασμένο, αν είναι τίμιο. Δεν πρόκειται δηλαδή να κάνω ανάλυση των ποδοσφαιρικών του προτιμήσεων. Εμείς λοιπόν είμαστε εκείνοι που πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερκεράσουμε την υποκρισία, να μην είμαστε προκατηλημένοι, αλλά να κρίνουμε έναν άνθρωπο κάτω από το πρίσμα των προσόντων. Όλα αυτά είναι σε αντίθεση με αυτά που είπαν οι προραλήσαντες. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι, όπως σας είπα, πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί. μάλλον τοποθέτηση εκφράσατε ή θέλετε να σας απαντήσει και στις έμεσες ερωτήσεις περί ποδοσφαιρικών προτιμήσεων. Βέβαια, καλά, ε, αστείευόμενος το είπα αυτό. Ναι, πέστε μας, πέστε μας ε, για ποιον είστε, ποιον στηρίζετε, τη Real Madrid ή τη γιατί αυτό ξέρετε μπορεί τελικά να είναι το καθοριστικό σημείο. Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσετε στην ερώτηση αυτή, αλλά αν θέλετε μπορείτε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επιφυλάσσομαι λέγοντάς σας ότι να, τα, παιδιά μου, τα παιδιά μου έχουν, προσυμπαθούν περισσότερο το, τη, τη λευκή φανέλα της Ρεάλ. Τέλος πάντων, προβληματιζόμενος πάνω σε αυτό όσον αφορά δηλαδή ε, την συμμετοχή και την εκπροσώπηση κάποιου αμερόληπτου οργάνου που έχουμε τέτοια στην Ισπανία, ακριβώ όπω ορίζει και η Συνθήκη τη Ένωση. Ε, τα, τα συντάγματα τη κάθε χώρα τελικά αυτό το οποίο αποδεικνύει την ανεξαρτησία στην άσκηση κάποιων αρμοδιοτήτων για κάποιο ανεξάρτητο όργανο, ε, τελικά αυτό αποδεικνύεται από τη διαδρομή, τη σταδιοδρομία, την παιδεία των μελών του οργάνου, και τον επαγγελματισμό τους και το καταστατικό φυσικά του θεσμικού οργάνου και εγώ στην ε, σταδιοδρομία μου πάντοτε έπρεπε να αναλάβω καθήκοντα που απαιτούσαν ε, ουδετερότητα γιατί ήμουν δημόσιος υπάλληλος. Και είμαι υπερήφανος ε, για το ότι η δημόσια διοίκηση της χώρας μου είναι ουδέτερη. Πέρασα δύσκολους διαγωνισμούς για να μπορέσω να γίνω επιθεωρητής των δημοσιονομικών. Τότε επί, επί Σολτσάγα ε, Υπουργεία Σοτσάγα στην Ισπανία. Και το Υπουργείο μου έδωσε αυτή την υποτροφία για να πάω για μεταπτυχιακά στην ΕΠΑ και ήταν σοσιαλιστής ο υπουργό τότε, ο κ. Σολτσάγα. Ε, αυτά που με ρωτήσατε, σας λέω. Όπως επίσης είμαι περήφανος για το ότι συνέβαλα και στην ε, ε, θέσπιση αυτού του εταιρικού φόρου. Ναι, το συλλογικό έργο ήταν τότε επί Σόλβες. Υπουργεία Σόλβες. Και εγώ ως υπάλληλο είχα υποχρέωση ουδετερότητας. Και εάν λοιπόν να λάβω καθήκοντα στο ελληνικό συνέδριο, βεβαίως και οι ικανότητέ μου θα μπουν στην υπηρεσία του Ελληνικού Συνεδρίου Συμφωνώ με τα ε, επιβαλόμενα ε, ανεξαρτησία, επαγγελματισμό κλπ. κλπ ό,τι ορίζει το καταστατικό. Ορτίθ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Κύριε υποψήφια, νομίζω ότι το βιογραφικό σας αποδεικνύει όλα αυτά που είπατε για τα προσόντα σας, την, ε, την ικανότητα κλπ. Πάντως, εμάς βασικά μας ενδιαφέρει το να είστε απολύτως ανεξάρτητος. Και γι' αυτό και έλαβα το λόγο να σας ρωτήσω, εσείς τι εγγύσεις παρέχετε για ανεξαρτησία όσον αφορά κάποια σφάλματα ε, όσον αφορά κάποια υποψηφιότητα. Κοιτάξτε, λέει ο υποψήφιο, ω μέλο του Ελληνικού Συνεδρίου, η δέσμευσή μου, η υποχρέωσή μου, το καθήκον μου είναι τον ενεργό συμφώνως με τους θεσμούς και τη συνθήκη της Ένωσης και να ενεργώ με απόλυτη ουδετερότητα χωρίς καμία παρέκκληση σε σχέση με χώρες ή θεσμικά όργανα. Αν λοιπόν συντρέξουν κάποια ασφάλματα, κάποιες παραβάσεις από πλευράς της χώρας μου, ε, θα πρέπει να ενεργήσω όπως θα ενεργούσα για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Βεβαίως και υπάρχει περίπτωση συγκρούσεως ε, συμφερόντων αλλά ε, ευτυχώ είναι συλλογικό το έργο στο ελληνικό συνέδριο, οπότε με διάφορο τρόπο θα γίνει, θα ρυθμιστεί αυτό. Εγώ πάντως θα δεσμευτώ όσον αφορά τους θεσμούς, την ε, λειτουργία και τη συνθήκη. Όπως ξέρετε, κανείς δεσμεύεται να τα τηρήσει όλα αυτά ενόρκως. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκάιερ. Από την δική μου πλευρά, λοιπόν, πρώτα μία παρατήρηση σχετικά με τη συζήτηση και προς τους κυρίους Οντί και Ριβελίνη. Ας τηρούμε ωστόσο κάποια συνέπεια στην γραμμή που ακολουθούμε. Και υπενθυμίζω ότι στη συζήτηση για την πρώτη πρόταση της Ισπανικής κυβερνήσεως προ λίγων εβδομάδων δεν αμφισβητήθηκε εν ουδεμιά περίπτωση η τεχνική κατάρτιση του υποψηφίου, τουλάχιστον από την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος. Διερωτήθηκαν εάν ήταν νόμιμη η υποψηφιότητα, διότι στο μεταξύ είχε αλλάξει η κυβέρνηση. Εγώ διαπιστώνω ότι εκείνη η υποψηφιότητα ε, ήταν απολύτως ε, νόμιμη όπως και τούτη εδώ. Και είχε αντιδράσει η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού στην ιδέα να μην συζητηθεί τα εκείνη διότι στο μεταξύ είχε αλλάξει η κυβέρνηση. Και διορτηθήκαν ορισμένοι μήπως ήταν και κομμουνιστής κατάσκοπος. Λοιπόν, οι τεχνικές, η εμπειρία του και οι τεχνικές του γνώσεις δεν είχαν αμφισβητηθεί καθόλου. Η ερώτησή μου τώρα ακολουθεί αυτή της κυρίας Ορτής. Στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού έχουμε το πρόβλημα ότι διαπιστώνουμε υψηλά ποσοστά ασφαλμάτων. Μήπως, επειδή, μήπως εδώ που μιλώ σας ενοχλώ, λέει ο, λέει ο κύριος Γκάιερ, πρόεδρος. Ναι, βρισκόμαστε σε... στην φάση της υποβολής των ερωτήσεων. Η αξιολόγηση θα γίνει μετά και οι πολιτικές τοποθετήσεις θα γίνουν in camera, δηλαδή και κλεισμένο των θυρών. Τώρα είναι μόνο η ώρα της υποβολής των ερωτήσεων. Ο κ. Γκάιερ. Ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, λοιπόν, διαπιστώνουμε υψηλά ποσοστά σφαλμάτων στην εκτέλεση του ε, κοινοτικού προπολογισμού και θέλουμε να τα μειώσουμε. Και εδώ μας χρειάζεται η συνεργασία των χωρών μελών που πολύ συχνά δεν είναι επαρκής. Το Ισπανικό Βασίλειο δυστυχώς είναι από τις χώρες εκείνες το οποίο με συνέχεια δείχνει πολλά σφάλματα στην διαχείριση των διαθωτικών ταμείων. Εγώ έχω κατανοήσει ότι πρόκειται εν μέρη διότι είναι πάρα πολύ περίπλοκη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ κεντρικής κυβερνήσεως στη Μαδρίτη και περιφερειακών κυβερνήσεων. Το κατανοώ αυτό, αλλά δεν απαλλάσσει το Ισπανικό κράτος, κράτος συγγνώμη, από το χρέος να μειώσει, από την υποχρέωση να μειώσει το ποσοστό. Κύριε Τομέ, να χρειαστεί να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Και υπάρχουν βέβαια κάποιες διατάξεις του καταστατικού του ελεκτικού συνεδρίου που ε, διασφαλίζουν την εξαρτησία του οργάνου αυτού, αλλά θα χρειαστεί να δεχθείτε να εγκρίνετε ορισμένες εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και να τις συνυπογράψετε και ίσως να μην είναι ιδιαίτερα θετικές και ωστόσο, για τη χώρα σας δηλαδή, και, ωστόσο θα πρέπει να τις υπογράψετε. πώς ε, θα είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα θελήσετε να παρέμβετε στις εκθέσεις αυτές. ποια θα είναι λοιπόν η συνεισφορά σας ως μέλους του ελεγκτικού συνεδρίου για την προσπάθεια μείωσης των σφαλμάτων στο Ισπανικό Βασίλειο. Πρόεδρος, επειδή περνά η ώρα, παρακαλώ όλοι να τηρείτε το όριο χρόνο αγορεύσεως και σας δίνω τον λόγο για να απαντήσετε σε αυτή τη σημαντική ερώτηση. Η υποχρέωσή μου ως μέλους του Ελληνικού Συνεδρίου είναι και έναν της Ισπανίας ίδια όπως και έναν των άλλων χωρών. Αν επομένως αναγύψουν κάποια σφάλματα αντικανονικότητες, όπως είδα και στο παρελθόν από πλευράς της Ισπανίας, όσον αφορά την διαχείριση των πόρων, στα πλαίσια των πολυπλόκων σχετικών διαδικασιών. Όλα αυτά θα επισημανθούν διόντως. Το θέμα είναι να μπορεί να ε, κάνουμε το καθήκον μας όχι μόνο στα, στα πλαίσια του προπολογισμού της Ένωσης όπου έχουμε τα σχετικά λάθη και επισημαίνονται κάθε χρόνο σε σχέση με την χορήγηση του, του, του πράσινου φωτός για την ε, του το ok για την ε, απαλλαγή για τον προπολογισμό. Ε, το θέμα είναι αυτό να γίνεται όποτε προκύπτουν τα λάθη. Θα πρέπει να βελτιώνει τη διαχείριση. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στους ελέγχους. Και εσωτερικά στα πλαίσια της Επιτροπής, αλλά και όσον αφορά τους εξωτερικούς ε, οικονομικούς ελέγχους ως προς τα κράτη-μέλη και όσον αφορά την σχετική απλούστευση των διαδικασιών Ήδη τώρα η συζήτηση που είναι τα δημοσιονομικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως έλεγε και στην πρώτη μου εισήγηση. Έχουμε τώρα μια πάρα πολύ εξαιρετική οικονομική συγκυρία λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης οπότε ε, είναι ακόμα πιο πολύτιμα από ποτέ τα χρήματα της Ένωσης. όλοι στο Ελληνικό Συνέδριο προέρχονται από κάποια χώρα. Ο καθένα έχει το δικό του προφίλ κλπ. Όμω ε, η ανεξαρτησία είναι δεδομένη και δεσμευόμαστε μόνο έναντι του θεσμικού αυτού οργάνου και δεν υπάρχει κανένα είδου οπισθοβουλία, επιφύλαξη σε σχέση με τη χώρα καταγωγή ή με άλλη χώρα. Σαν μέλο του Ελληνικού Συνεδρίου, αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να γίνεται η σωστή διαχείριση των χρημάτων τη Ένωση. Άλλωστε αυτό, αυτό θέλω και αυτό είναι το συμφέρον μου να γίνεται ως ισπανό πολιτή μέσα στου δύσκολου αυτού τους Η Ισπανική κυβέρνηση τώρα προσπαθεί να βάλει ένα καινούργιο δημοσιονομικό πλαίσιο σε συντονισμό με τις ε, διοικητικέ αυτόνομες περιφέρειες και τι τοπικές αρχές. Ούτω ώστε να υπάρχουν ε, ιδιαίτερα αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου κλπ. Ούτως ώστε να μην έχουμε σφάλματα, ε, λάθη ε, αντικανονικότητες σε σχέση με την ε, εκτέλεση κοινωνικών πολιτικών ή για άλλο λόγο. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και για την τήρηση του χρόνου. Ο κύριος Κυρακάκης. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε, για την παρουσίαση της υποψηφιότητάς σας. Είδα το βιογραφικό σας που είναι εξαιρετικό. Η πραγματική ερώτηση, κατά τη γνώμη μου, είναι πόσο ανεξάρτητος θα είστε απέναντι στο κόμμα σας, διότι είναι σημαντική σταδιοδρομία σας μέσα στο κόμμα σας, κάτι το οποίο δεν είναι κακό από μόνο του, αλλά επιτρέψτε μου να σας θέσω τρεις εξειδικευμένες ερωτήσεις και σας παρακαλώ απαντήστε μας όσο καλύτερα μπορείτε διότι πραγματικά προσπαθούμε, θα προσπαθήσω δηλαδή να αξιολογήσω και να καταλήξω στην ε, θέση μου στη βάση των απαντήσεων αυτών. Πρώτη λοιπόν ερώτηση, στην μακρά σας σταδιοδρομία ελεγκτού είχατε τυχαία την περίπτωση να αποκαλύψετε κάποια υπόθεση στην οποία συμμετείχαν μέλη του κόμματός σας ή αξιωματούχοι του κόμματός σας. Σε κάποια επίσης δεύτερον υπόθεση αρχής διαφωνήσατε δημοσίως με την κομματική γραμμή σας. Τρίτο, μπορείτε να μας αναφέρετε μία περίπτωση στην πολιτική σας ε, σταδιοδρομία όπου θεωρήσατε ότι η πίστη σας προς το κόμμα σας ερχόταν σε αντίθεση με το δημόσιο, δημόσιο χρέος σας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που ε, τηρήσατε το χρόνο αγορέσεως. Και σας παρακαλώ κύριε υποψήφιο απαντήστε. Ο υποψήφιος. Αυτό που ρωτήσατε αφορά το τι θα πει κανείς να είναι μέσα σε μια δημοκρατία μέλος ενός κόμματος όπου έχουμε πολίτες που εκφράζονται σε αυτή την κοινωνία μέσω αυτού του κόμματος. Και μιλούμε για βουλευτές, μιλούμε για μέλη πολιτικών κομμάτων. Αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν σε διαφορετικές ιδιότητες διαφορετικές κομματικές προτιμήσεις των μελών του Ελληνικού συνεδρίου. Εγώ είμαι μέλος του Λαϊκού Κόμματος εδώ και μία δωδεκαετία, αν δεν κάνω λάθος. Από το 2000. Αλλά και ο παδός, όλη μου τη ζωή. Φυσικά και υπάρχουν συγκρούσεις. Ε, συνέχεια. Πάντοτε τα όργανα ενεργούν συλλογικά. Όχι, όχι, δεν έχω συγκρουστεί με την ηγεσία του κόμματός μου, από ό,τι θυμάμαι. Να τώρα να αναφέρεστε σε κάποιο σκάνδαλο, σε κάποια περίπτωση διαφθοράς, κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν, ε, κάτι το οποίο έχει στιγματίσει κάποιο μέλος του κόμματος. Όχι, όχι, δεν είχα αντιμετωπίσει στην ε, διαδρομή μου αυτή κάτι τέτοιο. Όχι δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοια διλήμματα όπως αυτά που αναφέρατε. Και όπως άλλωστε λέει και το ερωματολόγιο, αν υπήρχε κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ένδικη διαφορά που να επηρέασε κάπως τη διαδρομή, η απάντηση είναι επίσης αρνητική. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και τώρα κιόλα ε, που είμαι ε, βουλευτής, εδώ και μια δεκαετία δεν ασχολούμαι με τη διαχείριση των δημοσιονομικών. Οπότε η ανεξαρτησία αποδεικνύεται κάθε μέρα στην άσκηση των καθηκόντων που έχει αναλάβει κάποιος. Δεν ξέρω, ελπίζω, κατάλαβα την ε, ερώτησή σας. Ελπίζω ότι σας καλύπτει η απάντησή μου. Ιδάλλως, αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, ευχαρίστω να σας την ε, παράσχω. Με Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόμέ. Ε, μια σύντομη συμπληρωματική είναι. Κύριε Σκυλακάκη. Δεν πρόκειται ακριβώ για συμπληρωματική ερώτηση. Απαντήσατε στις δύο πρώτες. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε και την τρίτη, θα την επαναλάβω. Μπορείτε να αναφέρετε μία σημαντική περίπτωση όπου θεωρήσατε στην κομματική σας σταδιοδρομία ότι η πίστη προς το κόμμα ερχόταν αντίθετη με τις ε, δημόσιες υποχρεώσεις σας. Όχι. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια τέτοια σύγκρουση κατά την οποία ως υπουργό, ως βουλευτής ε, και εκπροσωπώντας το κόμμα μου τέλος πάντων ότι ήρθα σε τέτοιου είδους σύγκρουση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου. Δεν, θυμάμαι, δεν θυμάμαι τέτοιου είδους προσωπική σύγκρουση συμφέροντα. Βέβαια, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι πολύ τάραχη η εσωτερική λειτουργία των κομμάτων. Κάθε φορά κανείς καλύτερα να τοποθετηθεί το πρακτέο. Σας ευχαριστώ. Μένουν τρεις ακόμη γραμμένοι συνάδελφοι. Ο κ. Μιλντερ πρώτα. Κύριε Μιλντερ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι στην απάντηση που δώσατε κύριε υποψήφιε γραπτός και την ε, επαναλάβατε και προφορικά ας υποθέσουμε ότι η παρούσα επιτροπή απορρίψει την υποψηφιότητά σας. Στην περίπτωση αυτή λέτε θα ζητήσετε από την Ισπανική κυβέρνηση να επανεξετάσει τον διορισμό σας. Αυτό το βρίσκω απολύτως ορθό. Αλλά ποια θα είναι η συνέπεια. Α υποθέσουμε ότι η Ισπανική κυβέρνηση θα πει όποια και αν είναι η γνώμη τη επιτροπή Ελέγχου προπολογισμού και ανεξαρτήτως αυτή, εμείς θα σα διορίσουμε. Διότι σύμφωνα με τη συνθήκη μπορούν να το πράξουν. Εσείς θα προχωρήσετε να αναλάβετε το καθήκον αυτό, γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και τελικώ και η Ολομέλεια θα είναι κατά τη υποψηφιότητά σα θα μπορέσετε να λειτουργήσετε παρά την αρνητική γνωμοδότηση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μπορέσετε να λειτουργήσετε ως μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ κύριε Μιούλτερ για την ε, ερώτησή σας. Κύριε Τομέ. Εγώ ψήφιος. Νομίζω ότι αυτό ξεκαθαρίστηκε στο ερωτηματολόγιο, διότι κατά τη γνώμη μου ε, το έργο το οποίο επιτελεί το ελεκτικό συνέδριο είναι έργο ε, απολύτου ανεξαρτησία, όπως ακριβώς ορίζει η συνθήκη και Πρόκειται για τεχνικό, τεχνοκρατικό όργανο. Έχει ε, βεβαίω ε, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν πολιτικέ αρμοδιότητε και ο έλεγχο γίνεται όσον αφορά την, τον προπολογισμό. Υπάρχει έλεγχο από εσά και από την Κομισιόν. Οπότε τελικά οδηγούμεθα κάθε φορά στην διαδικασία της απαλλαγής και αυτό γίνεται ε, με την λήψη της σχετικής απόφασης επί τη βάση της ετησίας εκθέσεως του Ελληνικού Συνεδρίου. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη λειτουργία είναι τα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου να απολάβουν εμπιστοσύνη από πλευράς της δικής σας Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Και όταν ορίζει η συνθήκη ότι αποφασίζει το Συμβούλιο και ε, αφού ακούσει το Κοινοβούλιο ή αυτό είναι ένας κανόνας, είναι μια διάταξη πολύ ουσιαστική που κάθε φορά θα καλείστε να συνεργαστείτε με το, με το δικαστήριο, με το ελληνικό συνέδριο, συγγνώμη. Νομίζω ότι στο ερωτολόγιο απήντησα ξεκάθαρα και θα ζητούσα από την κυβέρνησή μου να προβεί σε επιλογή υποψηφίου με συγκεκριμένα προσόντα τα οποία να προκαλούν την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ακολουθεί και αντεστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Γκρόνα γκρουπεν είναι bekymrad över hur enkelt det är för pengar från den... Ευχαριστώ λοιπόν. Η στην πολιτική μου ομάδα ανησυχούμε ιδιαίτερα για την παραοικονομία και τις απάτες που ασκούνται μέσω της παράνομης δραστηριότητας και των φορολογικών παραδείσων. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πώς, πώς χάνονται τα χρήματα αυτά από, μέσα από τους φορολογικούς παραδείσους. Sí, eh, el, el, el Tribunal de Cuentas Υποψήφιο, ναι. Το ελεγκτικό συνέδριο ως όργανο οικονομικού ελέγχου εξωτερικού και ανεξαρτήτου εκτελεί τα καθήκοντά του και ε, βεβαίω μπορεί να επισημάνει κάποια απάτη. Τότε επικοινωνεί με την Όλαφ ή τέλος πάντων με, όποια φορέα, με όποια αρχή είναι αρμόδια. Και από τη δραστηριότητά μας πηγάζουν συστάσεις και διάφορα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην βελτίωση της διαχείρισης και την καταστολή της απάτης. Και για το ΦΠΑ, όποτε γίνονται κινήσεις, χειραγωγήσεις, όσον αφορά την καταβολή, την ίσπραξη του ΦΠΑ σε κάποιες συναλλαγές διασυνοριακές, ναι, ναι, ναι έχουν, ε, έχει ε, ασχοληθεί με τέτοιε περιπτώσεις το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα, όσον αφορά τους του παραδείσους, κατά τη γνώμη μου, εδώ έχουμε μια πληγή και έχω εγώ προϊστορία, έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των καθηκόντων μου ως βουλευτού της χώρας μου. και ως προς αυτά συμφωνούμε με την αριστερή πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Πάντως, θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώνεται η διαχείριση σε όλα τα κρατημέλη και όσον αφορά τη λειτουργία των ε, ε, θεσμικών οργανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει ευρύτερη, ευρύτατη συνένεση, ακόμα και σε επίπεδο G20 για αυτά τα θέματα. Πριν από μια τριετία είχε γίνει μια συνάντηση στο Λονδίνο. Κάναμε και κάποια μικρά βήματα, αλλά συμφωνώ μαζί σα πρόκειται για κάποια πληγή όσον αφορά ε, την ε, χρήση των ε, φορολογικών παραδείσων για να παρακαμφθεί το δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τελευταία τον λόγο στην εισηγήτρια κυρία Γιάλα Σέντερ. Κύριε Σέντρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έγινε αυτή η συζήτηση όπως συνήθως γίνεται για τα θέματα τα οποία εγώ αναλαμβάνω σε Τέλος πάντων, ακριβώς αυτό το οποίο ήθελα ε, είναι να λάβουμε υπόψη αυτή τη μοναδική σύσταση της συνθήκης όσον αφορά τις ε, συνθήκες και προϋποθέσεις για τους υποψηφίους του Ελληνικού Συνεδρίου. Ακριβώς αυτό το οποίο ε, ζητείτε είναι η ανεξαρτησία. Όντως και ο Προκάτοχος και εσείς ε, επαγγελματικότατα ε, τα προσόντα σας είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά άλλα βέβαια τα πανεπιστημιακά, άλλα τα πολιτικά. Το θέμα είναι βέβαια το ότι για πρώτη φορά έκανε τέτοιο πράγμα μια κυβέρνηση. Και όλοι, όχι μόνο εγώ, εξεπλάγιμε. Και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με την εξαρτησία που έχετε. Κάτι το οποίο το απαιτούμε από όλους τους υποψηφίους. Γι' αυτό και ακριβώ και αυτά τα οποία λέμε εδώ δεν τα λέμε πάντοτε σε όλου του άλλου υποψηφίου. Λάβαμε υπόψη αυτά τα οποία είπατε. Πώ ε, διαχειριστήκατε το πρόγραμμα Ρέδε και επίση τι κάνατε ε, στα πλαίσια τη πολιτική σα σταδιοδρομία. Κύριε Μουγκρούθα, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο ακόμα εκρεμεί. Σημαντικό για μας. Γλώσσες. Για πέστε μας, εάν θα μπορούσατε να απαντήσετε στις ενδεχόμενες ερωτήσεις που σας απευθύνουμε σε κάποια άλλη γλώσσα. Μια που υπάρχουν συνάλφοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ισπανικά και πολλές φορές για να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία πέραν της διερμηνίας ε, πολλές φορές μιλούμε στα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου σε κάποια άλλη γλώσσα επομένως ε, πέραν της ισπανικής. Για πετε μας τώρα τι γίνεται με αυτά τα σφάλματα, αυτά τα οποία μας ε, προγραμματίζουν όλους όσον αφορά την ε, άσκηση της διαρκή πολιτικής. Ξέρετε, τα σφάλματα αυτά δεν ε, αφορούν συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν θέλαμε να κατηγορήσουμε κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά ε, γενικά μιλούσαμε για την περίοδο αυτή που ασχοληθήκατε και πώς μας απαντήσατε για την περίοδο 2000-2006. Αν έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Είναι συλλογικό όργανο το Συνέδριο. Τι γίνεται σε με το DAS για την απαλλαγή τι γίνεται με κάποια σημαντικά σφάλματα τα οποία έχουν βρεθεί ε, και στη Βαλένθια και στην Ανταλουσία. Πολύ σημαντικά. Και φυσικά αφορά και, και τα δύο μεγάλα κόμματα της κυβέρνησης και των δύο μεγάλων κομμάτων στην Ισπανία. Βεβαίως και προέρχονται από πάσα παράταξη τα μέλη του ελληνικού συνεδρίου Βεβαίως όμως και εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ικανή και ας μην είναι τόσο πολιτική όσο πανεπιστημιακή. Όντω πρόκειται για τεχνοκρατικό, τεχνικό ε, όργανο, αλλά πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη και την πολιτική προέλευση. Και είπατε ότι εάν λάβετε τη θέση αυτή. Είπατε ότι θα, θα είναι η δέσμευσή σας σαφής ε, και η συμμορφωσή σας με τα όσα επιτάσσει το, το δικαστήριο. Ο πρόεδρος στα αγγλικά. Παρακαλώ αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αρκετά φορτωμένη η μυρίσια διαταξή μας. Έχουμε τώρα τρεις ερωτήσεις από την εισηγητριά μας και επιθυμώ να τονίσω μία ερώτηση, να επισημάνω μία ερώτηση που έθεσε τα διαρθωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής είναι στις πρώτες προτεραιότητες ολόκληρως της ε, Επιτροπής και τα θέματα μας ενδιαφέρει να επιληθούν όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και αλλού. Τελευταία λοιπόν απάντηση παρακαλώ του υποψηφίου. Έχετε το λόγο. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Γνωρίζω ότι ως μέλος του, ελεγκτικού, ε, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν θα είναι απαραίτητα η γλώσσα εργασία μου τα ισπανικά. Έχω ενημερωθεί ότι υπάρχουν συνεδριάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που συνήθως διεξάγονται στα γαλλικά, αγγλικά ή γερμανικά. Δυστυχώς τα γαλλικά μου δεν είναι σπουδαία και δεν ομιλώ τα γερμανικά. Αλλά νομίζω ότι είμαι σε θέση να εργάζομαι καθημερινά στην αγγλική γλώσσα ε, για να διεξάγω τις εργασίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Βέβαια, τα αγγλικά δεν ήταν ποτέ η γλώσσα της καθημερινής μου εργασίας. Ελπίζω όμως ότι μπορώ να το βελτιώσω, μπορώ να τα βελτιώσω. Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά ζητήματα που θέτεται σχετικά με την δήλωση εξοπιστίας, της δυσκολίες που σημειώνονται στην Ισπανία, οι αυτόνομες ε, περιφέρειες στην Ισπανία και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τα διορθωτικά ταμεία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα θεωρώ ότι υπάρχει απολύτως καμία διαφορά σε μία διαδικασία ε, απέναντι στην Ισπανία ή απέναντι ε, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Εάν υπάρχει η αντίποτε αμφιβολία θα θέσω, για οποιοδήποτε θέμα δηλαδή, θα το θέσω υπόψη του ελεγκτικού συνεδρίου. Και άλλωστε το καταστατικό του δικαστηρίου, του ελεγκτικού συνεδρίου δηλαδή, είναι απόλυτα σαφές εν προκειμένου. Με... Μου ζητήσατε να αυτοπροσδιοριστώ ως πανεπιστημιακός, τεχνικός ή πολιτικός. Είναι δύσκολο για μένα να το πράξω αυτό. Άρχισα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία ως ε, δημόσιος υπάλληλο. Κατά κάποιο τρόπο εξακολουθώ να είμαι. Ποτέ δεν είχα ε, ιδιωτικό εισόδημα δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανάμειξη του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ε, στη δική μου περίπτωση δεν λέω αν αυτό είναι καλό ή κακό πάντως η ε, δέσμευσή μου ήταν πάντοτε στον δημόσιο τομέα ως δημόσιος υπάλληλο λοιπόν και σε υψηλές ε, θέσεις στην Ισπανική Διοίκηση αλλά και ως μέλος του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Για ένα διάστημα επίσης ήμουν ε, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης ε, για θέματα δημοσιονομικά στην Universidad Complutense της Μαδρίτης και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την περίοδο αυτή της επαγγελματικής μου ε, ζωής η οποία όμως διήρκεσε μόνο δύο έως τρία χρόνια ως επίκουρος καθηγητής. Όταν λέω πάντως ότι η δέσμευση των μελών στο Ελεκτικό συνέδριο είναι σημαντική, επιθυμώ να πω ότι γνωρίζω πολύ καλά το καθεστώς και τον κανονισμό που διέπειτα του ελεκτικού συνεδρίου και των μελών του. Τα γνωρίζω πολύ καλά. Και αυτό που μπορώ να συμβάλλω εγώ είναι η εμπειρία μου, οι γνώσεις μου, και η μελλοντική μου ανεξαρτησία που αυτή θα με διέπει καθημερινά στην εργασία του δικαστηρίου, βεβαίως στη βάση της ακεραιότητας της ανεξαρτησίας και του επαγγελματισμού που είναι οι βασικές εκείνες αξίες που έχει θεσπίσει το δικαστήριο για τις εργασίες του. Ο πρώτος. σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, διεξαγάγαμε μια εις βάθος ε, και εντατική ακρόαση και νομίζω ότι μπορώ να πω εξ ονόματος όλων των μελών της ε, Επιτροπής ότι θεωρούμε την δημόσια αυτή ακρόαση ως αναπόσπαστο μέρος μιας ε, ζωντανής δημοκρατικής ζωής. Ευχαριστούμε τον κύριο Τόμε Μπουκουρούσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που προσήλθατε. Ο υποψήφιος ευχαριστεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε και κλεισμένο των θυρών. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιος δεν ανήκει στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού να αποχωρήσει από την αίθουσα και να μπορέσουμε να αρχίσουμε αμέσως με το επόμενο στάδιο της ημερήσιας διαταξής μας.